Επίτροπε για τη συζήτηση. Ολοκληρώνεται η συζήτηση και ε, προχωρούμε στο επόμενο θέμα και θέλω να καλωσορίσω τον Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τον κύριο Φρανς Τίμερμανς, καθώς επίσης και την κυρία Υπουργό. Ε, δήλωση ε, Επιτροπής και Συμβουλίου για το κράτος δικαίου και τα θεμελιώδη δικαιώματα στην Ουγγαρία. Εξελίξεις από το Σεπτέμβριο του 2018 και μετά θα λάβει πρώτα το λόγο εξ ονόματος του Συμβουλίου η, κυρία Μελάνια Τσότ. Κυρία Υπουργέ, έχετε το λόγο, παρακαλώ. Κυρία Τσότ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αξιότιμη βουλευτέ, κύριε Επίτροπε, οι κοινέ αξίε όπω η ανθρωπινή αξιοπρέπεια, η ελευθερία, η δημοκρατία, η ισότητα, το κράτο δικαίου και τα ανθρώπινα δικαιώματα, είναι η η λύθη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και τα θεσμικά οργάνα αλλά και τα κράτη-μέλη θα πρέπει να σεβαστούν, να τις προστατεύσουν και να τις πρόθουν η Ρουμανική Προεδρία και όλοι μας. Συμφωνήσαμε ότι η προστασία του κράτους δικαίου, της δημοκρατίας και των ε, δικαιωμάτων είναι κάτι το θεμελιώδες για την Ένωση. Τις 18 Ενάτου του 18 το Συμβούλιο έλαβε ε, την τεκμηριωμένη γνωμοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 1. Ε, καλούσε το Συμβούλιο να καθορίσει και να διευνήσει κατά πόσον υπάρχει ε, παραβίαση ή κίνδυνος παραβίασης των θεμελιωδών αξιών υπό πλευράς της Ουγγαρίας και αυτό υποβλήθηκε τον Οκτώβριο, Νοέμβριο και Δεκέμβριο στο Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων. Στι 12 Ενδεκάτου το Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων έλαβε από την ε, Ουγγαρία μια έγγραφη απάντηση στην αιτιολογημένη πρόταση του Κοινοβουλίου και επίση μια παρέμβαση της Ευρωπαϊκή Επιτροπής όσον αφορά την εκκρεμούσα διαδικασία επί παραβιάση. κατά τη Ουγγαρία Το Δεκέμβριο οι Υπουργοί για πρώτη φορά αντίλαξαν απόψεις όσον αφορά τα επόμενα βήματα σύμφωνα με τη διαδικασία. Εμείς θα συνεχίσουμε την μελέτη και εξέταση αυτή τη αιτιολογημένη προτάσεω του Κοινοβουλίου. Δεν μπορούμε να προδικάσουμε, δεν μπορούμε να εξαγαγούμε συμπεράσματα όσον αφορά την κατάληξη της διαδικασία. Θα σα ενημερώνουμε όσον αφορά τις εξελίξεις μια που λαμβάνεται σοβαρά υπόψη ο προβληματισμός των ε, βουλευτών του Κοινοβουλίου και είναι κατακλείδη έχω να σας πω ότι τα θέματα τα οποία θέσατε κατά αυτήν την συζήτηση είναι κάτι κομβικό για την Ευρωπαϊκή Ένωση, για τη δική μας προσφύλωση αυτές τις αξίες, οπότε θεωρούμε ότι όλες οι πλευρές θα αντιδράσουν υπεύθυνα, τόσο ώστε να υπάρξει μια κατάληξη αυτής της διαδρομής σύμφωνη με τις ε, βασικές μας αξίες και σας ευχαριστώ. Εμείς ευχαριστούμε κυρία. Ευχαριστούμε κύριε Υπουργέ που μας παρουσιάσετε τη θέση του Συμβουλίου και τώρα ο Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο κ. Τίμερμαν. Ευχαριστώ το Κοινοβούλιο που προέβλεψε την κατάσταση της Ουγγαρίας σήμερα στην ημερήσια διάταξη. Η τελευταία φορά που συζητήσαμε την κατάσταση του κράτους δικαίου στην Ουγγαρία ήταν στις 11 Σεπτεμβρίου πέρσι. Την επόμενη μέρα το Κοινοβούλιο ανέκρινε το ψήφισμά του που ενεργοποιήσε το άρθρο 7.1 της συνθήκης και τη σχετικής διαδικασία κατά της Ουγγαρίας. Όπως έχω εξηγήσει και τότε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συμμερίζεται τι ανησυχίε ε, του Κοινοβουλίου όπω εκφράζονται στην ε, πρόταση που έχουμε μπροστά μα, ιδίω για τα θεμελιώδη δικαιώματα, ε, την προστασία του, τη μετακίνηση των Ρωμά και την ανεξαρτησία του δικαστικού κλάδου. Σήμερα θα ήθελα να σα ενημερώσω για τι πρόσφατε εξελίξει που έχουν λάβει χώρα από τον περασμένο Σεπτέμβριο, μεταξύ των οποίων των αποφάσεων του Συμβουλίου. Πρώτον, όπω έχω πει και το Σεπτέμβριο, σε αντίθεση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή βάσει της συνθήκης έχει ξεκινήσει η διαδικασία παραβάση και στην περίπτωση της Ουγγαρίας έχει ξεκινήσει πολλέ διαδικασίε παραβάσει που έχουν σχέση με τη αξία. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει αποφασίσει να χρησιμοποιήσει κατά το βέλτιστο δυνατό τρόπο την διαδικασία αυτή. Την περασμένη εβδομάδα στείλαμε μία επιστολή ε, σε σχέση με την νομοθεσία στο Ψόρο, η οποία επιβάλλει κυρώσει για διαδικασίε και αναστέλει αιτήσει ασύλου και αιτήσει διεθνού προστασία από οποιουσδήποτε είναι ύποπτη. Οι εγκρικέ αρχέ έχουν τώρα δύο μήνε να απαντήσουν στι κατηγορίε τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ιδάλω μπορεί να παραπέμψει την υπόθεση στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Επιτροπή. Επιπλέον, τον περασμένο Δεκέμβριο, το Ογκρικό Κοινοβουλίο ενέκρινε ένα νέο νόμο που ε, αναθεωρεί το εργατικό δίκαιο. Όπω ξέρετε, ο νέο αυτό νόμο έχει προκαλέσει έντονε διαδηλώσει στου δρόμου τη χώρα τι τελευταίε εβδομάδε. Αναλύσαμε την ε, συμβατότητα του νέου αυτού νόμου με την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία, ιδίω την ε, οδηγία για το χρόνο εργασία και αποστήλαμε σχετική επιστολή στι Ουγγρικέ Αρχέ. Βάσει τι απάντηση που θα λάβουμε, θα αποφασίσουμε για τα ενδεχόμενα μελλοντικά βήματα. Επίση, το Δεκέμβριο ακούσαμε ότι το Πανεπιστήμιο αν, της Κεντρικής Ευρώπης αναγκάστηκε να μετακινήσει την έδρα του από την Ουγγαρία στην Βιέννη. Το να έχουμε ένα πανεπιστήμιο που εξαναγκάζεται να φύγει από την Ευρωπαϊκή Ένωση λόγω κυβερνητικών μέτρων και συστηματικής πίεσης είναι άνευ προηγουμένου στην ιστορία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και είναι θλιβερό και πολύ ανησυχητικό να συμβαίνει κάτι τέτοιο στην Ευρωπαϊκή Ένωση παρά την διαδικασία που παραβάσει τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τι σαφεί προειδοποιήσει από πολλού ενδιαφερομένου και εταίρου. Ε, μια τελευταία εξέλιξη του Δεκεμβρίου είναι η συγχώνευση 400 ε, σταθμών μέσων μαζική ενημέρωση ε, που ελέγχονται από, από το κόμμα που είναι φιλεπροσκευμένο στην κυβέρνηση. Αυτό σχετίζεται και με την κυβερνητική απόφαση να εξαιρέσει την συγχώνευση αυτή από, την, από τον έλεγχο της αρμόδιας αρχής για τον ανταγωνισμό της χώρας και τον νόμο για τον έλεγχο των μέσων μαζική ενημέρωση. Στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, εξετάσαμε και τη λειτουργία του δικαστικού συστήματο στην Ουγγαρία, όπω την πρόθεση και τον τηρισμό των δικαστών, το πώ είναι οργανωμένη η εισαγγελία, και ε, το αν θα δημιουργηθούν νέα ε, δικαστήρια διοικητικού χαρακτήρα. Πέρσι τον ε, Δεκέμβριο το Κοινοβούλιο ενέκρινε δύο νόμους για την δημιουργία, την ίδρυση διοικητικών δικαστηρίων που θα αρχίσουν να λειτουργούν από το 2020. Είναι θλιβερό. Περιμένουμε τον Μάρτιο φέτος την έκθεση της Επιτροπής της Βενετίας για να δούμε τη συμβατότητα με το Ευρωπαϊκό Δίκαιο και τις Ευρωπαϊκές Προδιαγραφές. Η γνωμοδότηση της Επιτροπής της Βενετίας θα τροφοδοτήσει την τελική μας αξιολόγηση. Επιπλέον από τη διαδικασία υπεραβάση, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χρησιμοποιεί και άλλα μέσα, ελέγχους, έρευνες που έχουν να κάνουν με τη χρήση των ευρωπαϊκών κονδυλίων στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου και της ετήσιας διαδικασίας ε, δημοσιονομικών. Εκτιμούμε επίσης και τις συστάσεις προς την Ουγγαρία για να δούμε κατά πόσο καταπολεμείται η διαφθορά. Οι προσπάθειες για τη διαφάνεια, για τον ανταγωνισμό, ε, για τις δημόσιες συμβάσεις. Όσον αφορά τη διαδικασία του άρθρου 7. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δυστυχώς δεν έχει δώσει την ευκαιρία προς το παρόν ε, να περάσουν οι προτάσεις του στο Συμβούλιο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είπε ότι όποια και αν είναι η θέση τελικά του Συμβουλίου θα πρέπει να υπάρχει επεξεργασία της πρότασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου πλήρως. Αυτός είναι ο μόνος τρόπος και πρέπει να σέβονται αυτή τη διαδικασία όλα τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα. Θέλω να σας πληροφορήσω ότι τον Νοέμβριο, μετά από αίτημα της Αυστριακής Προεδρίας, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε στο Συμβούλιο μία επισκόπηση γεγονότων και δράσεων που έχει αναλάβει σε σχέση με την διαδικασία επιπαραβάση. Άσυλο, ε, βοήθεια προς τους ετούντες άσυλο, ανώτατη εκπαίδευση, διακρίσεις σε βάρος στο Ρώμα. Οι περισσότερες από αυτές τις περιπτώσεις εκκρεμούν ακόμα στο δικαστήριο. Όπως γνωρίζετε, η εγκρουγική κυβέρνηση ήδη απάντησε στην αιτιολογημένη γνωμοδότηση. Πιστεύω ότι το Συμβούλιο τώρα έχει όλα τα στοιχεία στη διάθεσή του προκειμένου να αρχίσει τη δικιά του αξιολόγηση των θεμάτων αυτών. Σας ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Ευχαριστούμε πολύ. Το λόγο έχει τώρα ο κύριος Τόμας Ντόιτς, εκ μέρους του ΕΛΚ. Ευχαριστώ. Γιατί η φιλελεύθερη πλειοψηφία για άλλη μια φορά βάζει το θέμα της Ουγγαρίας στην ημερήσια διάταξη, έτσι για να ακουστούν κάποιες ομιλίες ή γιατί με απελπισία προσπαθούν να τα βάλουν με την Ουγγαρία. Στην πραγματικότητα ο λόγος είναι ότι έρχονται ευρωεκλογέ και η αριστερή πτέρυγα, οι ε, φιλελεύθεροι θέλουν να τα βάλουν με την Ουγγαρία. Γιατί συμβαίνει αυτό όμως. Το γιατί συμβαίνει αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για την Ουγγαρία. Ουσιαστικά οι περισσότεροι στην Ουγγαρία συμφωνούν, ανεξάρτητα από ποιο κόμμα προέρχονται, ότι δεν θέλουν τη μετανάστευση. Οι περισσότεροι όμως εδώ θέλετε να στηρίξετε τη μετανάστευση, πιστεύετε ότι είναι ανθρώπινο δικαίωμα και θέλετε να νομιμοποιήσετε την παράνομη μετανάστευση. Θέλετε να σώσετε τα διάφορα προβλήματα και να τα λύσετε που έχουν να κάνουν με την ανάπτυξη μέσω από την παράνομη μετανάστευση. Θέλετε να αφαιρέσετε από τις χώρες μέλη το δικαίωμα που έχουν να προστατεύουν τα σύνορά τους ή για τις αποφάσεις τους σε σχέση με τις μη κυβερνητικέ ε, οργανώσεις. Ε, θέλετε, όπως και οι μη κυβερνητικέ οργανώσεις, ε, να εγκατασταθούν οι μετανάστες. Θέλετε εσείς να μας υπαγορεύετε πού θα εγκατασταθούν οι μετανάστες αυτοί. Θέλετε να μας τιμωρήσετε. Και ο κόσμος στην Ουγγαρία λέει όχι στη μετανάστευση. Εμεί όμω θα προστατεύσουμε τα σύνορά μα απέναντι στη μετανάστευση και με τον τρόπο αυτό προστατεύουμε και τα εξωτερικά σύνορα τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν θέλουμε να εισαχθεί το πρόβλημα στην Ευρώπη. Θέλουμε να εξαχθεί βοήθεια έξω από την Ευρώπη προς τις χώρες αυτές. Αυτό ζητούν οι Ουγγροί πολίτες. Γι' αυτό το λόγο εσείς έχετε πρόβλημα μαζί μας. Τέσσερις ε, μήνες πριν από τις εκλογές δεν εξυπηρετεί κανέναν απολύτως να επιτίθεστε κατά της Ουγγαρίας. Οι θα ψηφίσουν ώστε η Ευρώπη να αντιληφθεί επιτέλους το αυτό που πρέπει. Σας ευχαριστώ. Εξ ονόματος Σοσιαλιστών και Δημοκρατών, ο κύριος Βάιντεν Χόλσερ. Κύριε Πρόεδρε, με την εισαγωγή της διαδικασίας κατά της Ουγγαρίας έλαβε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μια σημαντική ιστορική απόφαση την οποία λάβαμε δύσκολα. Όμως μας επέκριναν πολύ διότι χρειαστήκαμε τόσο πολύ χρόνο. Ήταν αναγκαίο όμω αυτό διότι χρειάστηκε να συγκεντρώσουμε προσεκτικά όλες τις αναγκαίες πληροφορίες και βεβαίως να τις ζυγίσουμε υπεύθυνα. Το Κοινοβούλιο τον Σεπτέμβριο ψήφισε την έκθεση με σημαντική πλειοψηφία. Θα έπρεπε να περιμένει κανείς ότι μετά από αυτό θα ακολουθούσε μια κατάλληλη αντίδραση από πλευρά του Συμβουλίου Υπουργών και από πλευρά Ουγγαρία. Τίποτε τέτοιο δεν συνέβη. Η Ουγγρική κυβέρνηση, η οποία πριν δεν άφηνε καμία ευκαιρία που να μην εκμεταλλευτεί για να εμπλακεί στη διαδικασία, τώρα απεφάσισε να γνωρίσει το Κοινοβούλιο. Και η απουσία της σήμερα δείχνει την περιφρόνησή της προς το Κοινοβούλιο. Θεώρησε ότι δεν είναι υποχρεωμένη να λάβει υπόψη τις αμφιβολίες, τις, ε, την, των Ευρωπαίων φίλων της. Γιατί είμαστε φίλοι της. Η Ουγγαρία γίνεται όλο και περισσότερο μια δημοκρατία βιτρίνας. Δεσμεύει τα δικαστήρια, δεν επιτρέπει στις μη κρατικές οργανώσεις να λειτουργούν. Η πανεπιστημιακή ελευθερία βρίσκεται σε κίνδυνο και την πολιτική ανάλυση αντικαθιστούν πλέον θεωρίες συνωμοσία. Είναι εκπληκτικό το ότι το Συμβούλιο Υπουργών εξακολουθεί να μην λαμβάνει μέτρα για να ακολουθήσει αυτά που ζήτησε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Οι εξελίξεις, τις εξελίξεις τις λαμβάνει υπόψη σιωπηρά. Αυτό σημαίνει όμως ότι εγκαταλείπει την ιδέα της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Ελπίζω η Προεδρία του Συμβουλίου να μην καθυστερήσει περισσότερο για να λάβει τις τα αναγκαία μέτρα. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ αγαπητέ κύριε Βάιντεν Χόλτσερ. Θα δώσω τον λόγο τώρα στον κύριο Βίστισεν, εξ ονόματος της ομάδας συντηρητικών και μεταρρυθμιστών. Πάλι το Κοινοβούλιο ξεσπάει κατά της Ουγγαρίας για θέματα κράτους δικαίου και δημοκρατίας. Το ίδιο σώμα το οποίο πρότεινε να στερηθούν το δικαίωμα ταξιδιού άνθρωποι με του οποίου διαφωνεί. Το ίδιο σώμα, το οποίο εδώ στην Ολομέλεια πρόκειται να υπερψηφίσει τροπολογίες για τα άρθρα του κανονισμού, τα οποία στρέφονται κατά των απόψεων τη μειοψηφία στο ίδιο το Κοινοβούλιο. Αν δεν βλέπει κανεί αυτή την υποκρισία, τότε σημαίνει ότι έχει μείνει υπερβολικά πολύ μεγάλο διάστημα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Δεν γνωρίζω το ακριβέ περιεχόμενο των κατηγοριών κατά τη Ουγγαρία. Αυτό που γνωρίζω ωστόσο είναι ότι δεν υπάρχει ίση μεταχείριση των κρατών μελών. Βλέπουμε καταπίεση των διαδηλωτών στην Καταλωνία, βίαιη καταστολή των διαδηλώσεων, αλλά δεν βλέπουμε καμιά αντίδραση εδώ. Όταν υπάρχει καταστολή διαδηλώσεων στη Βουδαπέστη, προφανώ για το Κοινοβούλιο αυτό είναι παράβαση του κράτου δικαίου. Βρίσκω ότι είναι θεμελιωδώ προβληματικό. Ξεκινώντα από τον Γιώργ Χάιντερ στην Αυστρία πριν από 10 χρόνια μέχρι τι επιθέσει σήμερα κατά Ουγγαρία και Πολωνία, που ξεκινούν πάντοτε από το ευρωπαϊκό κατεστημένο. Και είναι βαθύτατα ενοχλητικό το γεγονός ότι εσείς εδώ δεν βλέπετε ότι το μόνο που κάνετε είναι να προκαλείτε ακόμα περισσότερη υποστήριξη για αυτούς που θέλετε να εξαφανίσετε, όπως τους Κατσίνσκι, Όρμπαν και λοιπούς και τους οποίους έχουν εκλέξει δημοκρατικά οι ευρωπαϊκοί λαοί. Τροπή για την Ευρώπη και τροπή για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ. Και τώρα η Judith της από τους Πράσινους. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πρέπει να καταλήξουμε ότι από την ε, ψηφοφορία της έκθεσής μου ε, το Σεπτέμβριο τα, τα πράγματα στην Ουγγαρία επιδεινώθηκαν. Οι Ούγγροι πολίτες έχουν κάθε λόγο να κατεβαίνουν στους δρόμους και πρέπει να τους δείξουμε λίγη. Θα ήθελα να σας απαριθμίσω μερικές από τις εξελίξεις του φθινοπόρου. Ο κύριος Τίμερμανς Επίσης αναφέρθηκε σε αυτά. Το Κεντρικό Πανεπιστήμιο αναγκάστηκε να πάει στη Βιέννη, γιατί η συμφωνία με... που, έχει υπογραφεί, που είχε συμφωνηθεί δεν θα υπογραφεί. Ε, ένα διοικητικό δικαστήριο δημιουργείται και το Υπουργείο Δικαιοσύνη είναι το αρμόδιο γι' αυτό. Ο πρώην Υπουργό τη Μακεδονία, ε, που έχει καταδικαστεί για διαφθορά, ε, προστατεύεται. 450 ε, ΜΜΕ ε, δημιούργησαν έναν όμιλο, έναν ενιαίο όμιλο με βάση νόμο. Επίσης, κάποια πράγματα που όλοι ξέρουμε, ότι οι Ούγγροι ε, χρονοτριβούν. Υποτίθεται ότι συνεργάζονται, μας κατακλείζουν με χαρτούρα, αλλά θέλουν να κερδίσουν χρόνο. Αυτό δεν μας εκπλήξει. Το γεγονός όμως ότι τα αιτήματα της Ρουμανικής ε, Προεδρίας να υπάρξει μόρφωση με το χνοδιάγραμμα είναι σαφές. Οι Ούγγροι πολίτε έχουν το δικαίωμα προστασία και πρέπει να ξέρουν ε, τι σκοπεύετε να κάνετε. Οι Ευρωπαίοι πολίτε πρέπει να ξέρουν τι θα κάνετε ε, και τι θα κάνουν οι πολιτικοί ηγέτε. Σα ρωτάω λοιπόν να λάβετε ευθύνη, να, να με καλέσετε στο Συμβούλιο και να αρχίσετε μια σοβαρή διαδικασία προς τους συναδέλφους ε, στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Ορισμένοι από εσάς είσαστε εδώ και χαίρομαι γι' αυτό, αλλά οι περισσότεροι δεν είστε. Συνεχίζω να σας εκτιμώ εσάς που υπερψηφίσατε την έκθεσή μου, αλλά έκτοτε τι κάνατε. Πού βρίσκονται οι ευθύνες σας, τις έχετε αναλάβει. Κυρία Σαρτζεντίνη, τελείωσε ο χρόνος σας. Μάλιστα και τώρα η κυρία Βεργιά έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Η Ουγγαρία είναι θαυμάσια χώρα, ε, ένα αμάλγαμα πολιτισμών. Ε, το σύμβολό της είναι η Βουλγαρία. Κανείς δεν θέλει να επιτεθεί στους Ουγγρούς πολίτες. Αλλά ο δικτά, δικτάτορας Ορμπάν θέλει να γίνει πρωταθλητής ενός ε, νέου μοντέλου εθνικιστικού και κατά των μεταναστών. Είναι κρίμα για την ιστορία αυτή τη όμορφη χώρα και τη Υπήρου μα. Από το Σεπτέμβριο ε, έχουμε τεράστιε διολυστήσει. Ε, διοικητικά δικαστήρια, ΜΜΕ που ε, και δικαστήρια που υποτίθεται κρίνουν δημόσια πράγματα είναι υπό ε, μεγάλη διαφθορά. Η Ουγγαρία δεν συμμετέχει στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Ε, μία νέα αυταρχική εισαγγελική διοίκηση δημιουργείται υπό τον Ορμπάν. Ε, υπάρχει ο νόμος ε, για τα εργατικά, ε, νόμος της σκλαβιάς όπως ε, λέγεται. Ο κύριος Τίμερμα, κύριε Τίμερμα, μάλλον τα ιδιολιστήσεις ξεκίνησε το 2010, παρακολουθείτε υποτίθεται τα πράγματα, εξετάζετε ποια είναι τα δικαιώματα. Δεν υπάρχει πόλεμος, λέω, στους Ούγκρους. Το θέμα των ε, μεταναστών είναι ε, ένα υποπροϊόν. Το βασικό είναι να σεβαστούμε τις αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ναι, όντως, χρονοτριβεί η Ουγγαρία πίσω από διαδικαστικά ε, έτσι, διαδικασίες, αλλά είναι προβληματική κατάσταση. Όλα Στούγκερ τώρα από, την, από το ΙΕΝΕΦ. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Στην Ολλανδία το 2014 37% ήταν η συμμετοχή στις εκλογές. Στην Ουγγαρία ήταν 70% για τις ε, εθνικές εκλογές. Και βγήκε ο Ορμπάν. Υπάρχει λοιπόν μεγάλη διαφορά στα ποσοστά με τα οποία ήρθαν εδώ οι ευρωβουλευτές, οι οποίοι ούτε καν στον ύπνο τους δεν βλέπουν τα ποσοστά της Ουγγαρίας. Αυτό πρέπει να το έχουμε υπόψη μας. Καθόμαστε και κάνουμε ψηφίσματα και ασχολιόμαστε με το Περού, τις εγκυμοσύνες, εκείνα κτλ. Μα δεν είναι σοβαρό αυτό. Οι Ευρωπαίοι πολίτες πρέπει να ενδιαφέρουν. Και αυτό ακριβώς κάνει και ο Ορμπάν. Ασχολείται με την ασφάλεια στη χώρα του. Και φροντίζει για τους ανθρώπους του. Και αυτή είναι η διαφορά. Ένας πρωθυπουργό ο οποίος ασχολείται με τον λαό του. Δεν είναι δυνατόν να βρίσκεται σε τέτοιες ε, διαδικασίες δικαστικές εις Το του. Άγαλμα θα έπρεπε να του είχαμε κάνει. Α φροντίσουμε λοιπόν να υπάρξει πρόβλεψη για τέτοιο κονδύλι στον προπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστούμε πολύ. Ο κύριος Παλτζότορα έχει το λόγο. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ αγαπητέ Πρόεδρε. Γίνεται αγώνας στη χώρα μου κατά της, δια, διαφθοράς και γι' αυτό ξεκινούν αυτά τα κηρύγματα μίσους. Είμαι πεπισμένος ότι αυτός ο πολιτικός αγώνας δεν μπορεί να συνεχιστεί εδώ στις Βρυξέλλες. Ο πολιτικός αγώνας πρέπει να γίνει στην Ουγγαρία μαζί με τους Ούγγρους πολίτες και πρέπει να χρησιμοποιήσουμε κάθε συνταγματικό μέσο για να ανατρέψουμε το καθεστώς Όρμπαν. Ευχαριστώ αγαπητέ συνάδελφε. Τώρα η κυρία Κούντριτσκα. Ευχαριστώ πολύ πρόεδρε. Ο νόμος είναι το μόνο μέσο που επιτρέπει σε ένα τόσο ποικιλόμορφο περιβάλλον όπως είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση να λειτουργεί. Όπως έλεγε η κυρία Στούσερ, είναι ακριβώς αυτό ο σεβιβασμός δηλαδή η ψυχή της δημοκρατίας. Αν όμως εμείς υπονομεύουμε τον νόμο και τις ευρωπαϊκές αξίες και αν δημιουργούμε έναν εναλλακτικό κόσμο προκειμένου να φέρουμε σε πέρα τους στόχους του δικού μας κόμματος, τότε έχουμε φτάσει στο τέλος της δημοκρατίας στην αρχή του τέλους. Δεν καταλαβαίνω γιατί οι Ουγγαροί συνάδελφοι δεν μπορούν να πείσουν τον ηγέτη τους ότι θα έπρεπε να προσπαθήσει να καταλήξει σε έναν συμβιβασμό και να υπάρχουν και πάλι οι βασικές αξίες της δημοκρατίας στην Ουγγαρία. Και έχω και μια ερώτηση. Δεν βλέπετε ότι δεν υπάρχει συμβιβασμός, αντίθετα υπάρχει κλιμάκωση της κατάστασης στην Ουγγαρία. Για παράδειγμα με την νομοθεσία για τα εργασιακά, το λεγόμενο νόμο της δουλείας ή ε, υποχρεώνοντας το Πανεπιστήμιο της Κεντρικής Ευρώπης να φύγει από τη χώρα. Είναι κοινικά αυτά, μα κάποιοι συνάδελφοι θα έπρεπε να έχουν δισταγμούς για όλα αυτά. Ευχαριστούμε. Σάνι τώρα εκ μέρους των Σοσιαλιστών. Ε, ευχαριστώ αγαπητέ Πρόεδρε. Προ τριακονταετίας έγινε μια σημαντική αλλαγή στην Ουγγαρία. Άνθρωποι που τότε είχαν συμβάλει στην αλλαγή αυτή είναι σήμερα ηλικιωμένοι, εύποροι και στην ουσία θεοδάρχες. Είχαν εκμεταλλευτεί το σοβιετικό σύστημα και τώρα, σήμερα δηλαδή, τα πράγματα είναι διαφορετικά. Έχει, μιλούμε για μια χώρα φτωχοποιημένη οι άνθρωποι στερούνται τα δικαιώματά τους, η γνώση έχει απαξιωθεί, η κατάσταση επιδεινώνεται διαρκώς. Οι εκπρόσωποι της εξουσίας και γενικότερα όλοι αυτοί που κυκλοφορούν με σωματοφύλακες εκπροσωπούν το έθνος. Μιλούν για πράκτορες, για πράκτορες του όρους, προσπαθούν να τους ανατρέψουν Αυτά είναι τα νέα από την χώρα μου, τη νέα χώρα της δουλείας. Ευχαριστώ. Κύριο Ζαβόρ. Ευχαριστώ. Ο Βίκτορ Όρμπαν δεν θέλησε να έλθει στην ε, συζήτηση, να προσέλθει στη συζήτηση. Έχει τα δικά του αυτός. Θα πρέπει ωστόσο γιατί θα χρειαζόταν τότε να προβάλλει επιχειρήματα αν ερχόταν δηλαδή. Εγώ τον ρωτώ τον Όρμπαν λοιπόν από εδώ. Τι είναι σημαντικότερο από το να συζητήσει με ποιον τρόπο μεταχειρίζεται και αντιμετωπίζει τις ευρωπαϊκές αξίες. Τι είναι πιο σημαντικό από το να συζητήσει ότι εδώ και εννέα χρόνια υπονομεύει τα δικαιώματα των Ούγγρων πολιτών στην Ουγγαρία. Η κατάσταση έχει επιδεινωθεί τα χρόνια αυτά. Έχει επιδεινωθεί σημαντικά. Στην Ουγγαρία συμβαίνουν πράγματα απαράδεκτα. Πρόκειται για ένα αυταρχικό σύστημα το οποίο έχει χαρακτηριστικά συστήματος Πούτιν. Τι πρέπει να γίνει επιτέλους ώστε τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα να λάβουν σοβαρά υπόψη τους την κατάσταση αυτή και να αντιληφθούν ποιο είναι ο κίνδυνο που απορρέει από αυτήν. Η κυρία Μπιόρκ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η κατάσταση δεν βελτιώνεται στην Ουγγαρία, αλλά βλέπουμε ότι ο Ορμπάν πιέζει περισσότερο όσου σκέφτονται διαφορετικά, είτε είναι ακαδημαϊκοί, είτε είναι μη κυβερνητικέ οργανώσεις, είτε άνθρωποι που υποστηρίζουν τα δικαιώματα των μεταναστών. Αλλά βλέπουμε ότι η αντίσταση στην κυβέρνηση επίση ενισχύεται πολύ στις χώρες μας, αλλά και εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το βλέπουμε αυτό και προσπαθούμε να αλλάξουμε την κατάσταση. Το Φιντές λέει ότι εγώ και άλλοι συνάδελφοι εδώ είμαστε εχθροί. Είμαστε αντίπαλοι, όπως και όσοι πιστεύουν σαν και εμάς στην Ουγγαρία. Αλλά κύριε Ορμπάν, όχι, δεν πρόκειται να εγκαταλείψουμε. Θέλουμε σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα, στο κράτος δικαίου, δεν θέλουμε τα δικά σας σχέδια εδώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση και θα συνεχίσουμε να υψώνουμε τη φωνή μας και να μιλάμε για τις ελευθερίες, για τα δικαιώματα των γυναικών, των μεταναστών και πράγματι θα είναι ένα από τα πιο σημαντικά θέματα για τις ευρωεκλογέ τις επερχόμενες. Βεβαίω, και εδώ θα στηρίζουμε πάντα τη δημοκρατία και το κράτος δικαίου. Ναι, θα είναι ένα θεμελιώδες ζήτημα, βασικότατο για τις ευρωεκλογέ γιατί τίποτα δεν είναι πιο σημαντικό από αυτό. Ευχαριστούμε κυρία Μουρβάη τώρα. Ευχαριστώ πολύ και ευχαριστώ την κυρία Σαρζεντίνη. Αλλά κυρία Σαρζεντίνη, για κοιτάξτε στην αίθουσα τι συμβαίνει, στην αίθουσα του ημικυκλίου. Γνωρίζετε ότι τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι 751. Ε, πάνω από μία δωδεκάδα δεν είναι παρόντα σήμερα και οι περισσότεροι είναι Ούγγροι. Βεβαίω τα πρόσωπα αυτά είναι εδώ, διότι η συζήτηση στρέφεται γύρω από την Ουγγαρία. Κατανοήστε επιτέλους ότι κανείς δεν ενδιαφέρεται για τον αγώνα που διεξάγεται κατά της Ουγγαρίας. Κοιτάξτε κυρία μου, τελείωσε ο αγώνας. Χάσατε. Ψάξτε να βρείτε κάποιο άλλο πράγμα να ασχοληθείτε. Και επειδή σας ενδιαφέρουν τα ανθρώπινα δικαιώματα, και εγώ άλλωστε ασχολούμαι με ανθρώπινα δικαιώματα, σας συνιστώ να κοιτάξετε με πιο βάρβαρο τρόπο καταστέλει η αστυνομία στην Γαλλία τις διαδηλώσεις. Δηλαδή γίνονται τα ίδια πράγματα όπως τότε παρημείνει στην Ουγγαρία πριν από το 2010. Άνθρωποι που έχουν χάσει την όρασή τους, έχουν υποστεί βαρύς τραυματισμούς στο κεφάλι και αυτά από τον αγαπημένο σας πολιτικό. Για ανθρώπους οι οποίοι ζητούν απλώς τα ανθρώπινα δικαιώματά τους. Να ασχοληθείτε και με αυτόν, κυρία Σαρτζεντίνη. Ευχαριστώ πολύ. είναι περισσότερα τα πρόσωπα που είναι παρόντα από αυτό που είπε η συνάδελφος. Κύριε Πρόεδρε, η κυρία Γκρέσλε, βρίσκομαι εδώ διότι ανησυχώ για λογαριασμό της ε, Επιτροπής Ελέγχου Προϋπολογισμού με το τι συμβαίνει με τα ευρωπαϊκά κονδύλια στην Ουγγαρία. Εμείς θεωρούσαμε ότι θα αυξηθεί το εισόδημα στη χώρα αυτή και θα μειωθούν οι άνεργοι. Δεν μπορούμε ωστόσο, το βλέπουμε αυτό, να προστατεύσουμε τα ε, ευρωπαϊκά κονδύλια όπως θα θέλαμε. Υπάρχει πρόβλημα διαφθοράς και υπάρχει πρόβλημα με δικαστικές αρχές οι οποίες δεν διώκουν ή δεν τους επιτρέπεται να διώκουν σχετικά εγκλήματα, ίσως διότι προστατεύουν κάποιους. Οι δημοσιονομικοί ελεγκτές έχουν άλλωστε πρόβλημα διότι η Ουγγρική κυβέρνηση δεν λαμβάνει απολύτω κανένα μέτρο για την καταστολή των περιπτώσεων αυτών. Κυρία Πρόεδρε του Συμβουλίου, σα παρακαλώ, φροντίστε ώστε να αρχίσει σύντομα τριμερής διάλογος όταν θα έχουμε τον σχετικό κανονισμό, διότι ο μετρητής διαφθοράς δείχνει την Ουγγαρία στον αριθμό 64, αμέσως μετά την Ελλάδα. Όμως στην Ελλάδα ο δείκτης κοιτάζει προς τα πάνω, δηλαδή τα πράγματα βελτιώνονται, ενώ στην Ουγγαρία όχι. Είμαι βεβαία ότι η Ουγγαρία μπορεί να τα καταφέρει και καλύτερα και θα ήταν πραγματικά ένα σημαντικό βήμα αποκατάσταση εμπιστοσύνη εάν αποφάσιζε η Ουγγαρία να συμμετάσχει στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Αγαπητέ Αντιπρόεδρε, κύριε Τίμερμαν, παρακαλώ να τα λάβετε σοβαρά υπόψη σα τα πράγματα αυτά. Σα ευχαριστώ που παρακολουθήσατε. Ευχαριστώ. Κύριε Γκρέσλε. Ο Ευχαριστώ. Ο Ούγγρος Πρωθυπουργό δήλωσε ότι σήμερα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο γίνεται μια συνεδρίαση σώρος και ότι πρόκειται για πολιτική φάρσα. Αυτά λέει η Ουγγρική κυβέρνηση. Με αυτόν τον τρόπο βλέπει η Ουγγρική κυβέρνηση την δημοκρατία. Ο Ούγγρος Πρωθυπουργό βεβαίω δεν είναι παρόν σήμερα εδώ, δεν θέλει να αντιμετωπίσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, διότι φοβάται τη δημοκρατία και φοβάται το δημοκρατικό διάλογο. Γι' αυτό και κατήργησε την ελευθερία του τύπου υπονομεύει την ανεξαρτησία τη δικαιοσύνη, δεν λαμβάνει μέτρα κατά τη διαφθορά η οποία έχει φτάσει και μέχρι τη δική του οικογένεια, δυσχεραίνει το έργο των οργανώσεων των δικαστών και προσπαθεί να στρέψει την χώρα προς δικτατορικέ κατευθύνσει. Δεν έρχεται στη Βραζιλία, πάει όμω. Δεν, συγγνώμη, δεν έρχεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν έρχεται εδώ στι Βρυξέλλε, πηγαίνει όμω στη Βραζιλία ή στη Ρωσία. Και προδίδει έτσι τα συμφέροντα τη ίδια του τη χώρα δεν μπορούμε να υποστηρίξουμε την πολιτική αυτή. Οφείλουμε να πούμε ευθαρσώ ότι αυτού του είδου η πολιτική δεν μπορεί να γίνει ανεκτή στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Κύριο Χάντσεν τώρα. Thank you, Mr. President. Ευχαριστώ. Αν ε, σήμερα ήταν να μπει η, Ευρωπαϊκή, η Ουγγαρία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν θα πληρώσει τα κριτήρια ένταξη Ε, ποινικοποιεί τους, ε, δεν δέχεται πρόσφυγες και ποινικοποιεί αυτούς που δέχονται ε, ε, τούντες άσυλο. Ε, εν τω μεταξύ κάποιοι άλλοι ε, λαμβάνουν την ε, ηθαγένεια όπως ο Ε, κυρίες και κύριοι, στον κατάλογο των ανθρωπίνων αξιών, ξέρετε πολύ καλά ότι οι Ούγγροι βρίσκονται πολύ χαμηλά γιατί υπάρχει τεράστια διαφθορά, όπως είπε η κυρία Σαρτζεντίνη και άλλοι. Ε, ζητήσαμε να σεβαστεί το κράτος δικαίου, αλλά εις Ε, η μείωση των πληρωμών προς τα κράτη, τα οποία δεν σέβονται το κράτος δικαίου, είναι σωστό ε, θέλω να πω στο Συμβούλιο πόσο πρέπει να περιμένουμε για να δράσετε, για να ενεργοποιηθεί το άρθρο 7. Θα πρέπει ε, να μην δείξουμε στενοχή ε, στην προσπάθεια ανατροπής του κράτους δικαίου. Ο Κάρλος Κοέγιο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι απλώς κοινή αγορά έχει κοινέ αξίες, αξίες που υπάρχουν και στην Χάρτα Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και στις συνθήκες. Όταν μιλήσαμε για τελευταία φορά για την Ουγγαρία, από τότε μέχρι σήμερα, εθνικοποίησε διάφορα ε, περιοδικά εφημερίδες, ραδιόφωνα, τηλεοράσεις ε, και αντιμετωπίζει με απάνθρωπο τρόπο τους πρόσφυγες. Η κυβέρνηση, ο πρόεδρος διακόπτη, γιατί υπάρχει πρόβλημα διερμηνίας ε, στα αγγλικά και στα πολωνικά. Και τώρα συνεχίζει ο κ. Σκουέγιο. Αποκαταστάθηκε το θέμα της διερμηνίας. Μήπως να ξαναρχίσω την παρέμβασή μου. Όχι, όχι, δεν χρειάζεται. Να συνεχίσετε από εκεί που είχατε σταματήσει. Λοιπόν, κύριε Πρόεδρε, εγώ θα ξαναρχίσω. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι μόνο κοινή αγορά. Έχει κοινέ αξίε, οι οποίε ε, σφραγίζονται και στην ε, χάρτα και στι συνθήκε. Από το Σεπτέμβριο, που μιλήσαμε τελευταία φορά, για τελευταία φορά για την Ουγγαρία, εθνικοποίησε η Ουγγρική κυβέρνηση τι περισσότερε ε, εφημερίδε, περιοδικά, ραδιόφωνα. Έκλεισε ένα πανεπιστήμιο φημώνει την αντιπολίτευση και αντιμετωπίζει απάνθρωπα τους πρόσφυγες. Η κυβέρνηση δημιουργεί κίνδυνο για το κράτος δικαίου ε, εις βάρος των Ούγγρων πολιτών και όλων των Ευρωπαίων πολιτών. Είναι μια κακή περίπτωση ο Ορμπάν ε, και υπάρχουν και άλλες χώρες, Πολωνία, Σλοβακία, Ρουμανία και Μάλτα που πρέπει να μας ανησυχήσουν και απασχολήσουν. Πρέπει να αντιδράσουμε, Πρόεδρε, πρέπει να δημιουργήσουμε ένα εργαλείο ελέγχου που θα αντιμετωπίζει ε, θέματα τέτοιες χώρες που δεν σέβονται τις, ε, τα ανθρώπινα δικαιώματα. Πρέπει να σεβόμαστε τις ε, θεμελιώδεις αξίες και θα πρέπει να πετύσουμε από το Συμβούλιο να ενεργοποιήσει το άρθρο 7 όπως προβλέπει η συνθήκη. Ελευθερία, δημοκρατία, κράτος δικαίου. Αυτές δεν είναι ηχηρές ε, λέξεις για να ξεκινάμε δεκάρικους λόγους. Είναι κομμάτια της ταυτότητάς μας η οποία απειλείται. Γι' αυτό ας έχουμε την, το κουράγιο να την υπερασπιστούμε. Ευχαριστώ. Ζητώ συγγνώμη για το πρόβλημα που υπήρχε και σας διέκοψα. Η κυρία Κίνγκα Γκάλ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κυρία Γκάλ. Όταν άκουσα τα όσα δήλωσε ο κύριος Νίντερ σκέφτηκα ότι είναι μάλλον αδιάφορο το τι κάνουμε, αφού δεν είναι παρόν ο Ούγγρος Πρωθυπουργό. Είναι όμω αυτό το πρόβλημα. Εγώ το βρίσκω γελίο. Όλοι και όλες γνωρίζουμε εδώ ότι η δράση αυτή είναι υποκειμενική και όχι αντικειμενική. Διότι αν αναλύσουμε τα πράγματα λεπτομερώς, θα έπρεπε να στραφούμε κατά όλων των χωρών μελών. Γνωρίζουμε ότι στην Ουγγαρία δεν έχουν κρατικοποιηθεί μέσα ενημέρωσης, δεν έχουν κλείσει πανεπιστήμια, τα πιστοποιημένα προγράμματα σπουδών στο Κεντρικό Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο εξακολουθούν να λειτουργούν. Πρόκειται για φάρσα δηλαδή αυτή η συζήτηση εδώ. Όλοι στρέφονται κατά της Ουγγαρίας, ενώ όλη αυτή η συζήτηση είναι μια αστεία παραγωγή, τα νήματα της οποίας κινούν κοινή αριστερά. Και όσοι είναι υπέρ της μετανάστευσης στρέφονται κατά της Ουγγαρίας, η οποία είναι αντίθετη με την υποδοχή μεταναστών. Η η κυρία Σαρτζεντίνη είπε ότι οι Ούγγροι πολίτες πρέπει να έχουν ακριβώ τα ίδια δικαιώματα όπως όλοι οι υπόλοιποι Ευρωπαίοι πολίτες. Αυτό σημαίνει ότι και οι Ευρωπαίοι πολίτες και οι Ούγγροι πολίτες έχουν το δικαίωμα να του αφήσει στη ησυχία του η κυρία Σαρτζεντίνη. Προχωρούμε στη διαδικασία Catch the Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε για άλλο ένα παράδειγμα της χρήσης διπλών μέτρων και σταθμών απέναντι σε ορισμένες χώρες μέλη. Το βλέπουμε αυτό διαρκώς. Επικρίνουν την Ουγγαρία για πράγματα τα οποία συμβαίνουν και σε άλλες χώρες μέλη και με τον ίδιο τρόπο. Όπως ο νόμος για τις υπερορίες ή η δικαιοδοσία των δικαστηρίων. Συχνά όμως ενημερώνουν με σφαλμένο τρόπο την κοινή γνώμη ή με υπερβολές ή κυκλοφορούν τα λεγόμενα fake news, οι ψευδεί ειδήσει. Δεν βοηθεί κανένα να διεξάγουμε τέτοιε απεραντοεπεί συζητήσεις γιατί δεν πάμε να δούμε τι γίνεται με τους Ούγκρους φοιτητές οι οποίοι δεν μπορούν τώρα να δώσουν εξετάσεις. Εδώ όμως διακυβεύεται η αξιοπιστία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Και δεν είναι δυνατόν να επικρίνεται διαρκώς η ίδια χώρα. Χουάν Λόπες Αγγιλάρη είναι ο επόμενος. Ευχαριστώ πρόεδρε, κύριε Αντιπρόεδρε Τίμερμανς. Για πρώτη φορά στην ιστορία μετά τη Λισαβόνα, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προχώρησε με τα δύο τρίτα πλειοψηφία στην πρωτοβουλία να ενεργοποιήσει το άρθρο 7 παράγραφο 1 σε σχέση με την Ουγγαρία. Και αυτό γιατί αυτά τα οποία περιγράφονται που κάνει ο Ορμπάν είναι μια κατάχρηση εξουσίας εντελώς ασύμβατη με τις αρχές και τις αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά του πλουμαρισμού κατά των μειονοτήτων, περιορισμός της ελευθερίας ε, ενημέρωσης αλλά και της ακαδημαϊκής ε, ελευθερίας. Και τα πράγματα χειροτερεύουν. Οπότε κύριε Τίμερμαντς, εγώ αυτό που θέλω είναι όταν αποφασίζει το Συμβούλιο παρουσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και συζητάει για τις συνέπειες μετά από την ψηφοφορία που με πλειοψηφία, όπως σας είπα, στα δύο τρίτα εγκρίθηκε ενεργοποίηση του άρθρου 7, θα έπρεπε τα τρία θεσμικά όργανα να ενώσουν τη φωνή τους και να πούνε φτάνει πια η κατάχρηση αυτή από την κυβέρνηση της Ουγγαρίας. Ευχαριστώ. Πρόεδρος, ευχαριστούμε πολύ. Τόμασιτς. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μια ένωση διαφορετικών χωρών με διαφορετικές παραδόσεις. Αυτό που μας συνδέει είναι κοινέ αξίες που δεν μπορούν βέβαια να παλύψουν τις διαφορές μας, ούτε τις διαφορές στην οτροπία μας. Ακριβώς επειδή έχουμε πολλές και διαφορετικές ε, λύσεις μπορούμε και προχωράμε. Ο συμβασμό είναι το βασικό, αλλιώ κάθε φορά η κάθε χώρα νιώθει ότι πλήττεται. Έχει μεγάλη παράδοση η Ουγγαρία και σίγουρα σκέφτεται διαφορετικά από ό,τι άλλε χώρε. Η Ουγγαρία αποφάσισαν για μια κυβέρνηση και η κυβέρνηση αυτή είναι απόλυτα νόμιμη και μπορεί κάλλιστα να επιλέγει το δικό της πρόγραμμα. Μπορούν να γίνουν ε, διαμαρτυρίες ειρηνικά για να εκφράσει ο κόσμος και αντιπολίτευση ε, την απόψή του και αυτό το επιτρέπει η κυβέρνηση και έτσι μπορούμε και εμείς και έχουμε διάλογο με την Ουγγρική κυβέρνηση. Οτιδήποτε άλλο είναι θέμα του Ουγγρικού λαού και η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν πρέπει να υπονομεύει τη δημοκρατία σε ένα κυρίαρχο κράτος. Ευχαριστούμε. Γιώργος Επιτίδιος τώρα, παρακαλώ. η ευρωπαϊκή ένωση κατηγορεί την ουγγρική κυβέρνηση ότι παραβιάζει τις αρχές του κράτους δικαίου και τα ανθρώπινα δικαιώματα ενώ για άλλες χώρες ανέχεται να συμπεριφέρονται με αυτόν τον τρόπο. ο πραγματικός λόγος για τον οποίο συμπεριφέρεται έτσι η ευρωπαϊκή ένωση είναι το ότι η ουγγαρία αρνείται να χορηγήσει πολιτικό άσυλο σε μετανάστες οι οποίοι διώκονται για ποινικά αδικήματα και σε άλλους οι οποίοι ελέγχονται και καθοδηγούνται από διεφθαρμένες ΜΚΟ. Αντί λοιπόν να συνεργαστεί με την ε, κυβέρνηση της Ουγγαρίας τόσο ώστε αυτή να χορηγήσει πολιτικό άσυλο στο ποσοστό και των μεταναστών που οφείλει να χορηγήσει, επιλέγει την οδό της συγκρούσεως. Όμως η κυβέρνηση της Ουγγαρίας προστατεύει τα συμφέροντα του Κρικού λαού. Δεν είναι σαν την ελληνική κυβέρνηση η οποία είναι ενδοτική ε, δέχεται και υποκύπτει στις πιέσεις και έχει μετατρέψει την Ελλάδα σε ένα απέραντο καταβλισμό δυστυχισμένων μεταναστών στους οποίους ούτε χορηγείται πολιτικό άσυλο ούτε τους δέχεται κάποια χώρα αλλά και ούτε απελάβνονται. Τελειώνω θέλοντας να πω ότι η συμπεριφορά αυτή προς την Ουγγαρία αποτελεί ε, το χαρακτηριστικό παράδειγμα της υποκρισίας της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Διότι ενώ στην Ουγγαρία συμπεριφέρεται έτσι, η Τουρκία αρνείται να ακολουθήσει την ίδια συμπεριφορά πρέπει να ολοκληρώσουμε πριν τα μεσάνυχτα την ε, Ολομέλεια σήμερα. Λέσλο Τόκας τώρα είναι επόμενος. Ευχαριστώ, ευχαριστώ πολύ αγαπητέ Πρόεδρε. Η απόψινή συζήτηση οφείλεται στους πράσινους και στους συνοδοιπόρους τους. Ήδη την τελευταία φορά που συζητήθηκε το θέμα εδώ, είχε καταδικαστεί η Ουγγρική κυβέρνηση. Πάλι καταδικάζεται η Ουγγαρία σήμερα, διότι η αριστερή και φιλελεύθεροι κάνουν στην ουσία ευρωπαϊκό προεκλογικό αγώνα εδώ. Και υφιστάμεθα εμείς το στίγμα στην Ουγγαρία οι χειρότεροι όμως είναι οι Ούγγροι βουλευτέ τη αντιπολίτευσης, οι οποίοι όπως και επί εποχής κομμουνιστικού καθεστώτος απεργάζονται την κατάρρευση της ένομης τάξη στην Ουγγαρία. Σας παρακαλώ να μην τους ακούτε. Ζήτω η Ουγγαρία, ζήτω η Ευρώπη. Ο κύριος το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι, κύριε Αντιπρόεδρε Τίμερμαντς, όταν γίνεται μια συζήτηση για τη δημοκρατία και το κράτος δικαίου στην Ευρώπη, εκείνος λέει «Α, συζητάτε μονίμως για την Πολωνία και την Ουγγαρία». Εγώ συμφωνώ λοιπόν με την ιδέα σας και ας ε, μιλήσουμε για την ε, ενεργοποίηση του άρθρου 7. Το κράτος δικαίου απειλείται αυτές τις μέρες από αυταρχικά καθεστώτα. Στην συνθήκη αναφέρεται ότι το άρθρο 7 μπορεί να ενεργοποιηθεί μετά από μία ψηφοφορία η οποία θα περάσει με τα δύο τρίτα των ψήφων των ψηφισάντων. Αυτό, δεν, αυτό το νούμερο δεν το φτάσαμε ποτέ το δύο τρίτα των ψηφισάντων. Στα αυταρχικά καθεστώτα, για να ξεκινήσει μια αντίστοιχη διαδικασία, ε, γίνεται νοθεία στις εκλογές. Πρέπει να σας πω το εξής. Ο Όρμπαν έκανε μία διάγνωση για το τι συμβαίνει σε αυτή την αίθουσα. Ευχαριστούμε πολύ. Τώρα το λόγο έχει ο Αντιπρόεδρος Τίμερμανς. Παρακαλώ. Ευχαριστώ. Να αντιδράσω σε κάποια από αυτά που άκουσα. Καταρχάς, αυτοί που λένε ότι δεν συμβαίνει τίποτα, είναι πολιτικό παιχνίδι εδώ, να σας παραπέμψω σε αυτά που είπα στην αρχική μου παρέμβαση. Ε, εμείς εξετάζουμε συγκεκριμένα πράγματα και θέτουμε ερωτήματα. Πιστεύουμε όταν πιστεύουμε ότι οι απαντήσεις σε αυτά τα ερωτήματα δεν συνάδουν με το ευρωπαϊκό δίκαιο, εμείς προχωρούμε. Έχουμε τον νόμο Stop Soros, να σταματήσουμε το σώρο. Η επανεγκατάσταση ε, εκτός της Ουγγαρίας ε, για το, το πρόγραμμα του, Ευρωπαϊκού, του Κεντρικού Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου. Κάτι έχει αλλάξει λοιπόν δραστικά και έχουμε ερωτήματα η συγχώνευση πάνω από 400 ΜΜΕ, χωρίς να μπορούν οι αρμόδιες αρχές να ελέγχουν αν αυτό συνάδει με την νομοθεσία. Όλα αυτά είναι συγκεκριμένα πράγματα. Η υιοθέτηση δύο νέων νόμων ε, για τα νέα ε, διοικητικά δικαστήρια. Συγκεκριμένο πράγμα. Ο νέος νόμος για τις υπερορίες. Έχουν συζητηθεί πολλά πράγματα σχετικά. Ερωτήματα γύρονται για το αν ε, συνάδει αυτό με το ευρωπαϊκό δίκαιο και την ευρωπαϊκή νομοθεσία. Και τώρα, ας πάμε στο θέμα αρχής που μπαίνει εδώ. Η δημοκρατία πάντα χρησιμοποιείται ως δικαιολογία για να μην συμμορφωθεί κανείς με την ευρωπαϊκή νομοθεσία. Αλλά δεν λειτουργεί έτσι η δημοκρατία, δεν λειτουργεί έτσι η Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ουγγαρία, ευτυχώς, Ε, επέλεξε, ευτυχώς επέλεξε, με κυρίαρχη απόφαση να γίνει μέλος τη Ευρωπαϊκής Ένωσης. Την ε, ενέκρινε το Κοινοβούλιο, επιβεβαιώθηκε από δημοψήφισμα του Ουγγρικού λαού. Αν αποφασίσει να γίνει μέλο μια οργάνωση που βασίζεται σε συνθήκε όπω η Ευρωπαϊκή Ένωση, λόγω τη επιλογή σου λε ότι θα ακολουθήσει του κανόνε τη συνθήκη. Και η Κομισιόν, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δηλαδή, έχει το καθήκον να εξετάσει εάν τα κράτη-μέλη ακολουθούν τους κανόνες της συνθήκης, οι οποίοι κανόνες είναι ξεκάθαροι για πολλά θέματα και ειδικά για το θέμα του κράτους δικαίου, άρθρο 2 και 19 της συνθήκης που λένε ξεκάθαρα για το διαχωρισμό των ε, εξουσιών, την ανεξαρτησία των μέσων ενημέρωσης κτλ. κτλ. Αυτά ψάχνουμε, αυτά κοιτάμε. Δεν θέλουμε να στυλιτεύσουμε χώρες που δεν θέλουν τους μετανάστες. Δεν θέλουμε να επιτεθούμε στην δημοκρατική λειτουργία ενός κράτους μέλους ή στην ε, πολιτιστική πολυμορφία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θέλουμε οι χώρες να λογοδοτούν για κάτι που επέλεξαν να κάνουν χωρίς να τις πιέσει κανένας. Ε, ελεύθερα έκαναν μια κυρίαρχη επιλογή. Επέλεξαν να ενταχθούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αυτή είναι η μορφιά της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης, ότι κάθε κράτος κυρίαρχα αποφασίζει. Ακριβώς γι' αυτό η Ουγγαρία επωφελήθηκε πάρα πολύ από αυτή την ένταξη. Και όλα τα άλλα κράτη-μέλη έδειξαν τεράστια αλληλεγγύη με την Ουγγαρία για να κλείσει το χάσμα και να εφημερούν οι πολίτες οι Ούγγροι όπως το αξίζουν. Αλλά δεν έχετε μόνο δικαιώματα Έχετε και υποχρεώσεις. Έχει υποχρεώσει η Ουγγαρία. Ε, υποχρεώσεις αναφέρονται στη συνθήκη και είναι καθήκον των Ευρωπαϊκών Θεσμικών Οργάνων, του Συμβουλίου, τη Ευρωπαϊκή Επιτροπής και του Κοινοβουλίου να φέρνουν, να ελέγχουν το πώς συμπεριφέρεται ο κανένα και να λογοδοτούν όλοι ενώπιον τους. Αυτό κάνουμε εμείς ενώπιον της Ουγγαρία. Τίποτα περισσότερο, τίποτα λιγότερο. Ευχαριστούμε πολύ. Κύριε Αντιπρόεδρε Τίμερμανς και τώρα η κυρία Τσότεκ μέρος του Συμβουλίου. Ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Αντιπρόεδρε, κυρίες και κύριοι, Σας διαβεβαιώ για άλλη μια φορά ότι η Προεδρία και το Συμβούλιο συνολικά δίνουν πολύ μεγάλη σημασία στην τήρηση του κράτους δικαίου και στην προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Είναι πράγματα τα οποία βρίσκονται στην καρδιά των όσων πιστεύουμε. Σας ενημερώνουμε για τις εξελίξεις και μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι η Προεδρία θα δώσει ιδιαίτερη προσοχή στις απόψεις που εκφράσατε σήμερα κατά τη διάρκεια αυτής της συζήτησης. Ακούσαμε τι ζητάτε και παραμένουμε ανοιχτοί υπέρ μιας πραγματιστικής προσέγγισης. Σας ευχαριστώ και πάλι για την προσοχή σας. Πρόεδρος, κυρία Χωτάλα στο Προεδρείο, ευχαριστούμε πάρα πολύ το Συμβούλιο. Και τώρα θα περάσουμε στο επόμενο θέμα